Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εκ νέου τις εργασίες της Επιτροπής μας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Σήμερα το απόγευμα, όπως ξέρετε, η Φιλανδία ανέλαβε την 1η Ιουλίου την Προεδρία του Συμβουλίου και είναι η πρώτη του τρίου των Προεδριών. Στη συνέχεια θα έχουμε την Κροατία το πρώτο εξάμεινο του 2020 και βεβαίως η Γερμανία, ε, τη Γερμανία από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του χρόνου. Είναι λοιπόν η πρώτη προεδρία αυτής της νέας ε, κοινοβουλευτικής περίοδου. Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα με μια ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου στους τομείς που είναι δική μας αρμοδιότητας, της Επιτροπής μας δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, όλες οι προεδρίες του Συμβουλίου αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικό φόρτο εργασίας. Όμως, ιδιαίτερα η δική σας αναλαμβάνει ακριβώς τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πρότασή μας για τις ε, τα νομοσχέδια, τις νέες νομοθετικές προτάσεις ε, στον τομέα της συνοχής και βεβαίως υπάρχει και η επιπρόσθετη δυσκολία που θα αντιμετωπίσετε με το Brexit που επίσης θα έχει αντίκτυπο στα ταμεία συνοχής. Στην φιλανδική, εκ μέρους της φιλανδικής κυβέρνησης, η υπουργό ε, Οικονομικών υπεύθυνη για ζητήματα συνοχής είναι εδώ μαζί μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά την κυρία Κάτρι Κολμούνη για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Νωρίτερα είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων χρήσιμη που μας επέτρεψε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, για την συνέχεια, για αυτό που μας περιμένει, δηλαδή την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων εν ώψη του γενικού κανονισμού, αλλά και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα συζητήσεων για τα άλλα ταμεία. Συζητήσαμε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν ε, τον, ε, το πολιτισμο πλαίσιο. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο την Υπουργό για μια πρώτη εισήγηση 15 λεπτών περίπου. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και στους ευρωβουλευτές σε δύο γύρους. Πρώτα στους συντονιστές και μετά τα μέλη της Επιτροπής μας. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και εκτιμώ που βρήκατε το χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη συνοχή. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα βλεπόμαστε συχνά κατά τη διάρκεια της Φιλονδικής Προεδρίας, αλλά και μετά από αυτή συνεχίζω ε, θα συνεχίσω να εργάζομαι εντατικά για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Χαίρομαι που έχω σήμερα αυτή την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας για τη Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η Φιλανδία έχει θέσει φιλόδοξο στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η πιο ανταγωνιστική και ε, κλιματικά ουδέτερη οικονομία παγκοσμία. Ο στόχο είναι κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, εμεί μαζί ω. Ε, νομοθέτες ε, να πετύχουμε ένα κοινό όραμα για μια νέα ε, στρατηγική ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία τη Φιλανδία, θεωρεί ότι τα κύρια στοιχεία θα περιλαμβάνουν τη μετάβαση προ μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, πραγματική ενία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, πραγματική ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια βιομηχανική πολιτική που θα διέπεται από την καινοτομία και τις ψηφιακές πολιτικές συμπεριλαμβανομένε, μια πολιτική εμπορική ενεργή ω εξωτερική διάσταση τη ανταγωνιστικότητα στις δεξιότητες και συνεχής μάθηση. Θα πρέπει οι κοινές μας προσπάθειες να μεταφράσουν αυτούς τους στόχους σε πραγματικότητα. Θα πρέπει η Ένωση να δράσει με έναν τρόπο που να παράγει αποτελέσματα ορατά στους πολίτες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι ότι ε, το νέο θεματολόγιο για την ανάπτυξη να παρέχει ένα πλαίσιο πολιτικής για τα επόμενα πέντε έτη. Ελπίζω ότι ε, την παραμονή πρωτοχρονιά ε, θα έχουμε έτοιμη μια τέτοια στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη για να εφαρμοστεί. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο λεπτομέρο στα πέντε στοιχεία που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο πολιτική για αυτό το θεματολόγιο ανάπτυξη, ξεκινώντα από το νούμερο 1, τη μετάβαση προ μια κλιματική κοινωνία. Το να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητο και είναι και οικονομική ευκαιρία, η έρευνα και η καινοτομία παίζουν σημαντικό ρόλο για να μετατρέψουμε αυτές τις ευκαιρίες ε, σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η μετάβαση ταυτόχρονα προς ε, μια τέτοια κλιματικά ουδετερή κοινωνία πρέπει να είναι δίκαιη, αλλά πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και νέα βιομηχανία. Ελπίζουμε ε, ότι δεν θα ταπανάτε τίποτα στο μέλλον. Επίσης, πολιτικές της ενιαίας αγοράς που θα βλέπουν προ το μέλλον και θα είναι εφοεί είναι σημαντικέ για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες, κυρίως ψηφιακές υπηρεσίες, ως ένα ολοκληρωμένο μέρος ε, της νέας αγοράς. Τρίτο, θα πω δύο λόγια για την σύγχρονη βιομηχανική πολιτική και την ψηφιακή οικονομία. Θα πρέπει να θέσουμε το στόχο η Ευρώπη να γίνει παγκόσμιο ηγέτη στην ψηφιακή οικονομία, ψηφιοποίηση ε, τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα και η οικονομία πλατφόρμας ε, είναι ε, παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμία αγορά τέταρτον. Οι νέες δεξιότητες και συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι απαραίτητε. Συνεχής μάθηση θα είναι στο επίκεντρο της επαγγελματικής ζωής στο μέλλον. Πέμπτον, η εμπορική πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο σε εξωτερική διάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υποστηρίζεται καλύτερα από φιλόδοξο ορθόδοξη εμπορική πολιτική που θα βασίζεται σε ανοιχτό πνεύμα και σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα. Αλλάζει η παγκοσμία τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να αποτελέσει έναν ισχυρό παγκοσμίο Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να συζητήσω το μέλλον ε, της, ε, των περιφερειών ε, και το επόμενο στάδιο της πολιτικής συνοχής. Ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των περιφερειών στο να οικοδομήσουν το μέλλον τους είναι κάτι σημαντικό για μένα, καθώς θεωρώ ότι η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ακόμα και της δικής μου περιφέρειας. Η πολιτική συνοχής συνεισφέρει σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και και σε όλε τι περιοχέ και μα βοηθά να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντικό εργαλείο ε, στο να προωθήσει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες, προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ανεργία, αντιγωνιστικότητα, δημογραφική αλλαγή, προσβασιμότητα και κλιματική αλλαγή είναι κοινέ σε όλα τα κράτη-μέλη και τις ε, περιφέρειες. Ταυτόχρονα, η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα, αποτελεσματική και να εστιάζεται σε θέματα. Η ενδυνάμωση των κοινών αξιών και του κράτου δικαίου είναι κύριε προτεραιότητε για την Προεδρία μα. Πρέπει να επικεντρώσουμε του κοινού μα στόχου που είναι σημαντική για το μέλλον τη Ένωση. Η χρηματοδότηση τη συνοχή μπορεί να φέρει τη θεμενή αξία για του πολίτε, βελτιώνοντα τι επενδύσει, την απασχόληση και την ευημερία. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να υποστηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινοτομία σε όλε τι περιφερειέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο στο να προχωρήσει την έρευνα και την καινοτομία και να δημιουργήσει ανθεκτικότητα στην παγκοσμιοποίηση. Ε, Τώρα, το να διερευνήσουμε ε, το δυναμική της ψηφιοποίησης σε νέες αναδυόμενες οικονομίες όπως η τεχνητή νομιοσύνη είναι σημαντικό για να έχουμε μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη και ορίζον Ευρώπη και οι πολιτικές συνοχή παίζουν σημαντικό ρόλο στο να προωθήσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Ε, Φύγει στρατηγικές εξειδικεύσεις αποτελούν καλό στρατηγικό πλαίσιο για την ε, οικονομική μεταμορφωσή των ευρωπαϊκών περιφερειών, επενδύσει σε τεχνολογίες με χαμηλή ενέργεια ανθρακά και λύσεις κυκλικής οικονομίας ε, σημειώνουν ένα σημαντικό ρόλο ε, αυξημένος στόχος για το κλίμα, δηλαδή δέσμευση του 25% για την πολιτική συνοχή είναι σημαντικό βήμα στο να υποστηρίξουμε αυτή τη στρατηγική. Επίση, ε, το να δώσουμε νέα προσόντα και να ενισχύσουμε τα προσόντα στην αγορά εργασία είναι σημαντική τομεί ε, στην ανταγωνιστικότητα, η ανάγκη για ισορροπένη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών και κοινωνικής ισότητας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη και δυνατή για να απαντήσει στις αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι επίση σημαντικό να ενδυναμώσουμε τη διασυνορική συνεργασία στα εσωτερικά αλλά και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κοινό συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθεί την κινητικότητα, τι επαφέ μεταξύ των ανθρώπων και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στι μεθοριακέ περιοχέ. Επίση, προγράμματα εξωτερικών συνόρων συνεισφέρουν στο να λειτουργούν και να είναι ασφαλή τα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, ουσιαστικά να διερευνήσει τι οικονομικέ ευκαιρίε που προσφέρονται από την περιοχή τη Αρκτική. Είναι ένα από του κύριου πρωταγωνιστέ στην Αρκτική και είναι προ το συμφέρον όλων των κρατών μελών να ενδυναμώσουν την παρουσία τη Ένωση στην περιοχή. Αυξημένε επενδύσει στην Αρκτική θα φέρουν προστιθέμενη αξία μέσω τη καινοτομία στον τομέα τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα βοηθήσουν την Ευρώπη να επιτύχει του στόχου τη Ατζέντα 2030. Το νομοθετικό πακέτο πολιτικής συνοχής 2021-2027 είναι σημαντική συνιστόσα του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία μας, σκοπεύουμε να προωθήσουμε το έργο αυτό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αγαπητά μέλη, η ολοκλήρωση του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι ένας από τους πιο σημαντικού πολιτικού στόχου κατά τη διάρκεια τη Φιλανδική Προεδρία το φθινόπωρο. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τι ε, διαπραγματεύσει. Επίση, θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε διάφορε ε, τομικέ προτάσει του πλαισίου. Σκοπεύουμε στο να έχουμε ένα ισορροπημένο πλαίσιο που να αντικατοπτρίζει τι νέε προτεραιότητε και τι παραδοσιακέ πολιτικέ. Επίση, πιστεύουμε ότι ένα ξεχρονισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει ε, να ανταποκρίνεται στι πολιτικέ προτεραιότητε τη Ένωση. Για την πολιτική συνοχή, η Προεδρία θα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τι διοργανικέ διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο αφού το Κοινοβούλιο θα έχει ξεκινήσει το έργο του. Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο να βρούμε μια κοινή συνεννόηση για θέματα που αφορούν ε, τον προγραμματισμό και το να ξεκινήσουν ε, σύντομα η επόμενη γενιά προγραμμάτων. Αν υπομονώ για επικοδομητική συνεργασία ε, μεταξύ των συνομαθητών για την πολιτική συνοχή. Δεσμεύομαι να προωθήσω το πακετό στο το περισσότερο κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να ολοκληρώσω τις παρατηρήσεις μου. Χρειάζεται η οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να είναι βιώσιμη περιβαλλοντικά και οικονομικά. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ένα νέο σχεδιασμό για την ανάπτυξη είναι απαραίτητο για τη μετάβαση προ μια κοινωνία κλιματικά ουδέτερη. Α θέσουμε αυτό το στόχο από κοινού, γεμάτη ελπίδα και φιλοδοξία και έτοιμοι να εργαστούμε. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι αντιγωνιστική και κοινωνικά να εντάχει σε όλους τους πολίτες απαντώντας στις προσδοκίες τους. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις και σχόλια. Είναι λοιπόν, μόνο για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Όπως προβλέπει η συνήθις διαδικασία, δίνω το λόγο πρώτα στους συντονιστές και μετά, εάν συμφωνεί και ο συνάδελφος Νόβακοφ, δίνω το λόγο πρώτα στον εκπρόσωπο των σοσιαλιστών, ο οποίος ε, θα χρειαστεί να αποχωρήσει κάποια στιγμή, ο κύριος Μάρκες. Και στη συνέχεια ο κύριος Νοβακοφ, αν δεν έχει εντύπωση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητέ κυρία Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή των Περιφερειακών Υποθέσεων. Ομιλώ εκ μέρους του συντονιστού μας. ήθελα να πω πως για μας το προσεχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζει ως κύρια πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, πολιτική συνοχή με την ε, προσθέμενη αξία που προσφέρει, με την αλληλεγγύη, με την, με την περιφερειακή συνοχή που προσφέρει στην Ευρώπη ολόκληρη και για λόγους πολιτικούς, γιατί έχει κρίσιμη σημασία και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. του του λεχθέντος. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τις θέσεις σας για αποτελεσματική χρήση των μέτρων. Ναι, πρέπει να υπάρχει η έννοια του κόστους και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Ταυτόχρονα να δούμε τις διαφορές μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και της ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνει ε, πολύ πιο απαιτητικέ ε, προβλέψεις για το προσοχές δουπού από αυτά που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη δεόντως και τις προτάσεις της Επιτροπής αλλά και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή την πολιτική της κοινής γεωργικής πολιτικής, τις λεγόμενες παραδοσιακές πολιτικές δηλαδή, που όμως έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την ευημερία των πολιτών, για τη συνοχή στην Ευρώπη και κυρίως για τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά και εν γέννη στα κράτη-μέλη, γιατί η πολιτική συνοχή είναι πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη. Ω τέτοια πρέπει να τη βλέπουμε και ω τέτοια πρέπει να τη, βλέπουμε, να τη θεωρούμε προτεραιότητα για το προσεχέ πολιτέ στο πλαίσιο. Προσδοκούμε λοιπόν να είναι κατάλληλο και προσαρμοσμένο στι ανάγκε και προσδοκίε των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πολιτές νοσονομικό πλαίσιο και πώ σα περιμένουμε τα αντίστοιχα. Υπάρχουν κάποιε προτεραιότητε που πρέπει να λάβουμε υπόψη την απανθρακοποίηση, πολύ μεγάλη προτεραιότητα και σημασία πολιτική, πρέπει να ενσωματωθεί στο Πουδουπού, ψηφιοποίηση που αναφέρατε και εσείς ως προτεραιότητα της Προεδρίας σας, που σημαίνει ότι πρέπει η καινοτομία να μπει σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προαγάγει και την καινοτομία, που επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των άκρως απομακρυσμένων περιοχών, ε, που χρειάζονται περισσότερο την αλληλεγγύη μας, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ισότιμες ευκαιρίες, άρα και αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα στο επόμενο πολιτές οικονομικό πλαίσιο. Και για να κλείσω κάποια λόγια για τις ε, περιοχές μέσου εισοδήματος Έχουμε δει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης να επιτρέψει την ανάπτυξη και την άνοδο ορισμένων περιφερειών, αλλά ορισμένες μπορεί να βρεθούν παγιδευμένες σε μια μέση θέση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι αναφέρεστε και σε αυτό. Βεβαίως δεν έχει κλείσει ο διάλογος με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, εξασφάλιση ποσών για τις περιοχές αυτές σε κάθε είδος πολιτικής και βεβαίως ακόμα έχει να γίνει πολλή συζήτηση για να γίνει ε, να ενσωματωθεί στο προσχέδιο σπουδουπού και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε, όπως είπαμε, μεγάλη πλειοψηφία ε, από το προηγούμενο κοινοβούλιο και που περιμένουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη με σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Νόβακοφ από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργή. Κυρία Υπουργέ, ε, εκ μέρου του ΕΛΚ δεν θα σα καλωσορίσω στην Επιτροπή μα, Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε συχνά το επόμενο εξάμεινο. Ε, ξέρετε, εσεί οι Φιλανδοί είστε διάσημοι, γνωστοί για τον ανοιχτό σα χαρακτήρα και την ε, ειλικρίνειά σας και θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ αυτό. Άκουσα το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας. Από τις 17 σελίδες η πολιτική συνοχή αναφέρεται μία φορά, σε μία παράγραφο. Και γίνεται μάλιστα αναφορά στην, στις περικοπές της πολιτικής συνοχής. Εγώ περίμενα κάτι περισσότερο. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές σας ε, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε ε, σε μια φάση διαπραγμάτευσης της επόμενης επταετούς περίοδου. Μπορείτε το Σεπτέμβριο ε, να προχωρήσετε τις διαπραγματεύσεις. Έχετε εντολή για να κλείσετε τουλάχιστον δύο ή τρία κεφάλαια διαπραγμάτευσης. Θεωρείτε ότι μπορούμε ε, να ε, επαναπροσδιορίσουμε ε, κάποια στοιχεία στην διαπραγμάτευση όπως το θέμα της χρηματοδότησης και το ποστός χρηματοδότησης σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Merci beaucoup, pour le groupe euh, Renew. Ευχαριστώ ο κύριος Καντέκ από το, την ομάδα Renew, ο κύριος Κνότεκ, συγγνώμη. Σας ακούσαμε με μεγάλη χαρά να αναφέρεστε στις προκλήσεις ε, ε της μετάβασης προς μια ε, Ευρώπη χωρίς άνθρακα. Αναφερθήκατε επίσης στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και πρέπει να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Νομίζω ότι συμφωνούμε και ως προς το ότι στις προτεραιότητές σας ε, δεν λέγονται πολλά για την πολιτική συνοχή. Θα ήταν καλό λοιπόν να γίνει κάτι και προς την κατεύθυνση αυτή. Μιας και είστε εδώ σήμερα, θα ήθελα με την ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα που αντιμετωπίζουν κάποιες περιφέρειες που έχουν ε, που επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την πρόκληση της ουδετερότητας ό,τι αφορά την εκπομπές άνθρακα. Ε, υπάρχουν δηλαδή ε, βιομηχανίες με εντατική χρήση άνθρακα, ε, που έχουν, έχει αυτός ο κλάδος ε, μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσει. Ε, θα υπάρξει υποστήριξη ε, προς αυτές τις περιοχές στο πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νένας για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ε, είπε μια φράση στα φιλανδικά ο μιλητής. Συγγνώμη, αυτά είναι τα φιλανδικά που ξέρω. Και από ό,τι ξέρουμε η φιλανδική διπλωματία είναι διάσημη και τη φέρατε μία από τις πιο σωστές μέρες του χρόνου έχουμε ένα από τα πιο καυτά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ω παγκόσμιοι παίκτε. Είναι η προβληματική τη κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό που ήδη στο πρόγραμμά σα είπατε ότι θέλετε να κάνετε κάτι σχετικά. Έτσι λοιπόν σας βλέπω περισσότερο σαν εταίρο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο ήταν σαφές ε, για την ε, μείωση του άνθρακα στη βιομηχανία και τα αποτελέσματα των εκλογών μας δείχνουν ότι και οι άνθρωποι, οι πολίτες το θέλουν αυτό. Θα σας ε, έλεγα λοιπόν, θα σας ρωτούσα αν ε, θα υιοθετήσετε τη θέση του Κοινοβουλίου για την μείωση του άνθρακα και την απαγόρευση σχετικά με τα ορεικτά καύσιμα. Τι θα κάνετε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις επίσης θέλετε, είπατε, να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσει στο φθινόπωρο. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ καλό στόχος, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βιαζόμαστε σε κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Αν τα καταφέρετε, εγώ θα χαιρόμουν να δεχτείτε την πρόταση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνετε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω Πώ ακριβώ θα διεκπαιρεώσετε την όλη διαδικασία, θα την κάνετε βιαστικά ή θα πάρετε χρόνο για να έχετε μια συνεκτική πολιτική συνοχής. Και φτάνω τώρα και σε ένα άλλο ερώτημα. Είπατε, η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω για την ισχύ τη. Αυτό είναι ένα από του πολλού λόγου που πρέπει να αυξήσουμε τι δαπάνε στην πολιτική συνοχή. Και όλοι οι προλαλήσαντε το είπαν αυτό. Θα ήθελα να πείτε ποια είναι η θέση της Προεδρίας του Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Αν μπορούμε να δούμε αύξηση, που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γράψατε στην ε, δήλωσή σας. Όταν ε, μιλάμε επίσης ε, για την αφαίρεση του άνθρακα, αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει μέσω, από τη, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Και μια τελευταία ερώτηση για σας. Είπατε ότι η περιοχή της Αρκτικής είναι πολύ σημαντική για σας. Ναι, φυσικά. Είναι και η γεωγραφία που παίζει ρόλο. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την περιοχή της Αρκτικής. Ναι, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή στην Αρκτική αν πρόκειται να σώσουμε την φύση στην Αρκτική, την περιοχή, τις θάλασσες αλλά και το βυθό της θάλασσας αλλά αν ε, τα σχέδιά σας ε, είναι παρόμοια με τους Ρώσους, δηλαδή απλώς να προβείτε εκεί σε εξόριξη πετρελαίου, αυτό είναι εντελώ ε, διαφορετικό και δεν θα πρέπει να εργαστούμε υπέρ αυτού. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ομάδα Ίντε. Αλεξάνδρο Πάντσα. Ή εσείς, κυρία μου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα την ε, εισήγησή σας και αισθάνομαι την υποχρέωση να σας επισημάνω τις ανάγκες και απαιτήσει και των περιφερειών της Νότιας Ευρώπης και κυρίως αυτές, αυτών που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είμαι ενήμερη βέβαια και για την ε, ιδιαίτερη προσοχή που θα δώσει η Προεδρία σας στο εξάμεινο αυτό για την ε, προαγωγή της γραφικής συνοχής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ότι αυτό αφορά πολλέ περιφέρειες και όχι μόνο την περιφέρεια της Αρκτικής. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αν θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή όπως χρειάζεται άλλωστε στις ε, ζώνες της Νότιας Ευρώπης από τις τελευταίες ε, έρευνες αποδεικνύεται ότι υπάρχουν περιφέρειες στην Ιταλία, όπως και η ιδιαίτερη μου πατρίδα η Σικελία, που καταγράφονται στις πιο στις ε, περιοχές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, για τον αλφαβητισμό, για τις υποδομές κυρίως. Και μετά όσα μας είπατε πολύ σωστά και επισημάνατε, όπως συνέπειες της κλιματικής αλλαγής κτλ. Θα ήθελα επιπλέον να συμπληρώσω υπογραμμίζοντας το ότι οι περιοχές της Μεσογείου ακριβώς είναι αυτές οι οποίες υφίστανται τις μεγαλύτερες ζημιές από την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας του πλανήτη, ιδιαίτερα στη Γεωργία που έχουμε τις μεγαλύτερες ε, ζημιές εμείς στις περιοχές μας λόγω των κακοκαιριών που προξενεί. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στα κονδύλια της σύνοχης όπως και της ανάπτυξης. Πάνω απ' όλα για τις υποδομές και δεν αναφέραμε μόνο στις ψηφιακές για τις οποίες οπωσδήποτε χρειάζεται αυτή η παρέμβαση που προβλέπετε αλλά και ε, εδαφικές υποδομές οι οποίες έχουν χαρακτήρα θεμελιώδη μπορούμε να τις εντάξουμε ακόμη και στην έννοια μιας ανοιχτής και προσβάσιμης πολιτικής για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης σε σχέση με την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το ψηφιακό θεματολόγιο στην πατρίδα μου και την περιοχή μου ήδη παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Και έτσι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη όθεση και στους νέους αλλά και στους λιγότερο νέους προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω λοιπόν να ληφθούν υπόψη αυτές οι ανάγκες στον προγραμματισμό σας για να ε, καλυφθούν επαρκώς και αυτοί οι τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. ECR. Φίτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση, τουλάχιστον όσον αφορά τις ενδείξεις που μας δώσατε, την εισήγησή σας. Τα θέματα που θίξατε φυσικά και τα μοιραζόμαστε είναι προτεραιότητες δράσης και θα πρέπει να τις υποστηρίξει όχι μόνο η δική σας η Προεδρία, αλλά γενικά η πολιτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να κάνουν με σημαντικούς τομείς ε, και ιδιαίτερα για το τομέα της συνοχής έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η συνοχή έχει πολύ, μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πρόγραμμα για τη συνοχή είναι πολύ φιλόδοξο, γι' αυτό και Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία και να δοθούν απαντήσεις στις ανάγκες. Πρέπει να εντοπιστούν, πιστεύω, ορισμένα ζητήματα στα οποία θα ήταν σκόπιμο και βέβαια με την ταχύτητα δράσης που επίσης επισημάνατε και την υποστηρίζουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δοθούν και κάποιες πιο τεχνικού χαρακτήρα απαντήσεις ε, γιατί και τις συμμερίζομαι στις αδρές γραμμές τους ε, της προσεγγίσης σας, θα ήθελα πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για να δούμε τι μας περιμένει σε αυτή την χρονική περίοδο που ακολουθεί και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην ταχύτητα δράσης μας σε σχέση με την ικανότητα ταχαίως προσδιορισμού των όρων με τους οποίους θα εξασφαλιστούν οι πόροι από το 2021 και μετά τι είδους χρονοδιαγράμματα, τι είδους συγκεκριμένε προτάσεις έχει υπόψη της η Φιλανδική Προεδρία. Η δεύτερη σκέψη έχει να κάνει με την ε, γραμμή που θα θέλατε ενδεχομένω να ακολουθήσετε σε σχέση με την ε, ανάκτηση ορισμένων δαπανών που δεν έχουν αξιοποιηθεί ε, ορθά και τρίτον θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν ζητήματα και ασυνέπεια στην πολιτική συνοχή, με την έννοια δηλαδή τη ευελιξίας. Βλέπουμε ότι καλούνται τα κράτη να χρησιμοποιούν εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας όμως και Ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει την δυνατότητά τους για συμμετοχή στη συνοχή. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν τα δικά μου τα ερωτήματα, πιο τεχνικά αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο να απαντηθούν για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε ώστε να επιδιώξουμε τους κύριους στόχους και τους κύριους άξονες της πολιτικής της Προεδρίας σας. Κλείνω και εγώ με μια επισήμανση σχετική με την ανάγκη στις περιφερειακές ζώνες να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε επίπεδο. Βεβαίως η περιοχή της Αρκτικής έχει τη μεγάλη σημασία που γνωρίζουμε όλοι, αλλά ταυτόχρονα για την εδαφική συνοχή ίσως θα πρέπει να δούμε και άλλες πτυχές της Ευρώπης. Και γι' αυτό είναι σημαντικό σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις και για τις άλλες περιφερειακές ζώνες της Ευρώπης, ώστε να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι στόχοι ή διαφορετικές εκτιμήσεις, ενδεχομένως πολιτικές ε, που θα αναγνώριζαν ε, ιδιαιτερότητες για αυτές τις περιφερειακές ζώνες ε, για τις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τις ε, επιπλέον δράσεις που θα αναπτυχθούν στο προσεχές διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κ. Παδημούλης, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Καλώς ορίζω, κυρία Υπουργέ. Ε, μας παρουσιάσατε σε αδρές γραμμές της απόψεις Φιλανδικής Προεδρίας για τα θέματα της συνοχής και του Γενικού Προϋπολογισμού, αλλά αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, οι αριθμοί δείχνουν ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι ανισότητες οι περιφερειακές στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί και έχουν αυξηθεί και οι κοινωνικές ανισότητες. Άρα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά για να ενισχύσουν τη συνοχή, διότι η πολιτική συνοχή σημαίνει μείωση των ανισοτήτων, όχι αύξηση των ανισοτήτων. Άρα, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτή είναι η θέση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ολομέλειάς του και όχι μόνο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, που είμαστε σήμερα εδώ, ότι θα πρέπει οι πολιτικές για τη συνοχή να ενισχυθούν και επομένως τα κονδύλια για την πολιτική συνοχή να ενισχυθούν και να μην μειωθούν. Έχουμε μια πρόταση της Κομισιόν η οποία οδηγεί σε μια μείωση μεσοσταθμική των κονδυλίων για τις πολιτικές συνοχής κατά 8%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αντίθετο και ζητάει να μην περικοπούν τα κονδύλια της συνοχής, αντίθετα να αυξηθούν. Εκτός από τον φιλόδοξο στόχο σας να καταλήξει σε συμφωνία το φθινόπωρο η Φιλανδική Προεδρία, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς σε ποια πλευρά στέκεστε, είσαστε υπέρ της μείωσης των κονδύλιων συνοχής ή υπέρ της διατήρησής του και της αύξησής του. Και θα ήθελα σε αυτό μια πιο συγκεκριμένη απάντηση από τη Φιλανδική Προεδρία. Επίσης, συμμερίζομαι το στόχο σας για να υπηρετηθεί η εδαφική συνοχή. Αλλά εκτός από το παράδειγμα της Αρκτικής που μας αναφέρατε, ενδιαφέρον και σωστό, υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Νότος. Υπάρχει και η νησιωτικότητα, η οποία στη χώρα μου την Ελλάδα περιλαμβάνει πάνω από 200 κατοικημένα νησιά. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στον Ευρωπαϊκό Βορρά και την Αρκτική, που είναι πιο κοντά στη χώρα σας διότι θα πρέπει η Προεδρία, η εκάστοτε Προεδρία να ενδιαφέρεται για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε υπάρχουν πολλοί Φιλανδοί και Φιλανδές που επισκέπτονται και τη χώρα μου και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Και το τελευταίο, επειδή υπάρχει στο Συμβούλιο μία διαμάχη ανάμεσα στις χώρες που είναι net contributors και net receivers σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Και αυτό οδηγεί σε συμβιβασμούς με τη μέθοδο του ελάχιστου κοινού παρανομαστή στο να μειώνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Υπάρχει μια πρόταση που λέει για να την ξεπεράσουμε αυτή την αντίθεση να αυξήσουμε τους ίδιους πόρους. Υπάρχουν οι προτάσει της Επιτροπής Μόντι, υπάρχουν προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λένε επειδή χρειαζόμαστε χρήματα για να υπηρετήσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας βρούμε και νέου ίδιου πόρου από τη φορολόγηση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τη φορολόγηση των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. Πώς βλέπει η Φιλανδική Προεδρία αυτές τις προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ. ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε μετά από αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές θα ζητήσω από σας να απαντήσετε στα ερωτήματα που τέθηκαν. Σημειώσατε, ε, θα διαπιστώσετε μάλλον τα ερωτήματα αυτά είναι πολλά, αλλά ότι συγκλίνουν τα ερωτήματα. Υπάρχει δηλαδή μια ανησυχία, μια πραγματική ανησυχία, σε σχέση με τις θέσεις του Συμβουλίου, υπάρχει μια απόρριψη, σαφής απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει και μια αποφασιστικότητα της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Θα πρέπει να διατεθούν δημοσιονομικά μέσα για την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά ή τουλάχιστον να διατηρηθούν. Και βεβαίως υπάρχουν και ανησυχίες σε σχέση με το ποσοστό της χρηματοδότησης που στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγεί σε μείωση. Οδηγείται σε μείωση. Υπάρχει δηλαδή εδώ μια προσμονή στο τι θα κάνει το Συμβούλιο. Εάν λοιπόν η συνοχή αποτελεί όντως προτεραιότητα για τη Φιλανδική Προεδρία, αναμένουμε ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα πρέπει να αφιερωθεί στο θέμα της συνοχής και αναμένουμε ως ήθιστε σε κάθε Προεδρία του Συμβουλίου να λάβει χώρα και μια άτυπη Υπουργική Σύνοδος αφιερωμένη στη συνοχή. Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό και τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε μεταξύ μας. Ε, αναμένουμε από εσά, ε, κυρία Υπουργέ, απαντήσεις, σαφείς απαντήσεις, σε ό,τι αφορά τη θέση του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό με τις κοινέ διατάξεις καθώς και βεβαίως να απαντήσετε και στα υπόλοιπα ερωτήματα που σας θέθηκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τα σχόλια όλους τους βουλευτές και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν καλύτερα και θα συνεχίσουμε βέβαια μετά τη συζήτηση. Όπως και να έχει ο στόχος της ε, Φιλανδικής Προεδρίας, θέλω να πω, είναι να εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοδότηση να μπορέσουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα αυτό και το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θέλω μια ισορροπία στο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις νέες προτεραιότητες, αλλά και τα παραδοσιακά στοιχεία και τους στόχους των πολιτικών. Οι Μάρκες Νόβα, να μίλησαν για το χρονοδιάγραμμα. Να σας εξηγήσω συγκεκριμένα τι σκοπεύουμε να κάνουμε και πώς. Το Συμβούλιο έχει μια μερική κοινή θέση για το Γενικό Κανονισμό. Η Φιλανδική Προεδρία είναι διατεθειμένη να ε, επανεκκινήσει τον τριμερή διάλογο για το πακέτο συνοχής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άπαξ και το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να αναλάβει δράση, πράγμα το οποίο αναμένουμε να δούμε κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και μπορώ συγκεκριμένα να πω πως ε, θα δώσουμε προτεραιότητα στο γενικό κανονισμό, ε, θα σπεύσουμε να προωθήσουμε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την προγραμματική περίοδο 2021 και μετά. Τα προγραμματικά χαρακτηριστικά βεβαίω και στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τη συνοχή, για την ευημερία των πολιτών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουν αυτέ οι συνομιλίε, κυρίω στα πιο ακανθώδη ζητήματα. Ε, ξέρω βεβαίω ότι υπάρχει ανάγκη να συζητηθεί και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, αλλά αφού θα έχει κλείσει πρώτα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τον κύριο Φίτο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζήτησε. Κοιτάξτε, το Συμβούλιο έχει μια μερική εντολή, η οποία στηρίζεται στο Γενικό Κανονισμό για τα διάφορα ταμεία και το Ιντερεκ. Έχουμε ξεκινήσει τις συνομιλίες με το Κοινοβούλιο σε πολιτικό επίπεδο, μάλλον και τεχνικό επίπεδο. Αυτό θα συνεχιστεί το ταχύτερο δυνατό, οι συνομιλίες με το Κοινοβούλιο. και κυρίως όσον αφορά και τον κανονισμό που είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπής απασχόληση Έρπλους. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συζητητέ του. Το ζήτημα της ε, διευθέτησης της μετάβασης, ε, έτσι ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο απρόσκοπτη η μετάβαση από τον προηγού στο προηγούμενο στο επόμενο προγραμματικό πλαίσιο είτε διοικητικά δηλαδή, είτε με τριμερείς διαλόγους, είτε με αιρεσιμότητες, με ζητήματα που θα αποσκοπούν σε αξιολόγηση αποτελεσμάτων, θα τα καταφέρουμε μέσα από τον τριμερή διάλογο αυτό. Επίσης, κανονισμοί αναθέματα για τα χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά ή το Interreg, ε, όλα αυτά είναι κεντρική σημασία θέματα. Επίσης, τι άλλο θα μπορούσα να πω σε σχέση με τις ερωτήσεις που άκουσα. Ναι, ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολούν είναι η κλιματική αλλαγή. Πώς δηλαδή μπορεί η πολιτική συνοχή να αποτελέσει εργαλείο για να απαλλαγούμε από τα ορυκτά ε, καύσιμα, παραδείγματι, και να, ανατρέψουμε, να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή η οποία τόσο επηρεάζει τις ζωές μας. Εδώ βρισκόμαστε στον πυρήνα της, ε, του σχεδιασμού μας, ε, του προγράμματος εργασίας μας Και εδώ θα ενταχθούν όλες οι κλιματικές προτεραιότητες. Η χρηματοδότηση αυξάνεται κατά 25% του, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για την κλιματική αλλαγή. Αυτό ξέρω ότι τη χάνει υποστήριξη. Για μας έχει σημασία η πολιτική συνοχή να προσαρμοστεί σε αυτό το στόχο. Άλλο στόχος της ε, πολιτικής συνοχής, το πρασίνισμα, το greening, ε, η καθαρή οικονομία, πιο πράσινη οικονομία και κυκλική οικονομία, κλιματικές αλλαγές, πρόληψη κινδύνων. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αρκετά φιλόδοξες προτάσεις σε σχέση με το ισχυρό πρόγραμμα. Επίσης, ε, ερωτήσεις άκουσα σε σχέση με τις περιφέρειες και την συμπερίληψη ή λήψη υπόψη καλύτερα όλων των περιφερειών. Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν και οι ε, άκρως απομακρυσμένες περιοχές, ε, οι υπερπόντιες περιοχές, οι πιο απομακρυσμένες, οι πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Και βεβαίως αναφέρθηκα εγώ στην Αρκτική στην ε, εισήγησή μου. Καθώς από πλευρά Φιλανδία αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε περιφέρεια είναι ε, ο τόπος κατοικίας ε, κάποιων ανθρώπων συγκεκριμένων, ένας τόπος ο οποίος μπορεί να έχει στοιχεία ευάλωτα, φύση ευάλωτη που πρέπει να προστατευθεί και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε και την απασχόληση και το ε, οικονομικό δυναμικό που υπάρχει στις περιοχές αυτές. Έγινε λόγος για τα ορυκτά καύσιμα. Ναι. Βεβαίως προσπαθούμε να αποσπαστούμε από αυτά. Αυτή όμως η επιλογή έχει συνεπεί σε όλες τις ε, περιφέρειες. Οι νησιωτικές, τα αρχιπέλαγα, η Μεσόγειος, οι παράκτιες, τα νησιά, όλα αυτά θα χρειαστούν κάποιες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες ε, διευθετήσεις, αφού έχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως τόποι διαβίωσης. Και αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δηλαδή αυτές τις ε, περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές, σε παραδείγματι. Η νομοθεσία για την περιφερειακή συνεργασία νομίζω ότι λαμβάνεται ε, γνήσια υπόψη από το Συμβούλιο ισότιμα για όλες τις περιφέρειες. Ε, επιπλέον θα μπορούσα να συμπληρώσω το εξής. Για τον ε, κύριο Πρόεδρο, για την ερώτηση στην πολιτική, το επίπεδο ε, λήψη αποφάσεων και συνεδριάσεων που οργανώνονται. Έχουμε λοιπόν άτυπη σύνοδο υπουργών για την συνοχή που δεν έλαβε αποφάσεις όπου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα με τον τριμερή διάλογο να προχωρήσουμε. Υπόθηκε επίσης ότι πρέπει το χέτερο δυνατό να προχωρήσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να οργανώσουμε ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τη συνοχή, ειδικά εάν αυτό μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου. Για τον κύριο Φίτο επίσης την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα και την πολιτική συνοχής αλλά και τη σταθερότητα, το, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα σημεία διαπραγμάτευσης. Και νομίζω ότι είναι όριμο για να περάσει και στον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ, ελπίζοντα ότι έχω δώσει απαντήσει σε όλε σα τι ερωτήσει. Ή τουλάχιστον έκανα ό,τι μπορούσα για να απαντήσω. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Συνάδελφος ο κύριος Αρήμου, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είπατε στην ομιλία σας ότι είναι σημαντικές για σας ε, οι ε, παραμεθόριες περιοχές και περιφέρειες ε, και ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν και για αυτές προτάσεις νομοθετικές και να προχωρήσουν γρήγορα. Στο τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η υπερσυνοριακή συνεργασία με το Interreg με 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως την επεξεργαστήκαμε, ε, αναφέρεται ε, σε 108 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για την επταετία και ερωτώ το εξής. Πολύ απλά. Εμείς στην Επιτροπή μας γνωμοδοτήσαμε προς την ίδια κατεύθυνση ομόφωνα σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής διεκδικώντας έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα αφορά ένα έτο ένα ποσό των 11 εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, δηλαδή ζητούμε περισσότερα από όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα και περισσότερα από όσα αυτή τη στιγμή διατίθενται για το Ιντερεκ και για το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Εσεί ω Φινλανδική Προεδρία θεωρείτε ότι μπορείτε να εισαγάγετε αυτή την απέτηση και να την υποστηρίξετε στο διάλογο στο Συμβούλιο και να υπερασπιστείτε τι ε, θέσει ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Αρκεί να μου πείτε ναι ή όχι. Merci. Ευχαριστούμε. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο. Έτσι λοιπόν θα σας παρακαλούσα να είστε σύντομοι. Η κυρία Νταμάτου, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Υπουργό που βρίσκεται εδώ. Διάβασα πολύ προσεκτικά το προγραμματικό έγγραφο και το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, κυρίως ε, η προσοχή που δίνεται στα περιβαλλοντικά. Είναι λογικό το ερώτημα λοιπόν. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερη πολιτική συνοχή. Ναι, όμως ε, ε, να υπάρχει και μια δράση αναχέτησης της ε, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει γίνεται σεβαστό το κράτο δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό βεβαίως ολόχης βάρος της πολιτικής συνοχής που βοηθά κυρίως τι λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Πολιτική Συνοχή ήδη έχει καθορίσει τη θέση του στις ε, κύριες εκθέσεις. Ε, μιλώ για τον κοινωνισμό περιοδικών διατάξεων, ε, για την εδαφική περιφερειακή συνεργασία και για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι και απευθύνουμε έκκληση προκειμένου η Προεδρία της Φιλανδίας να χωριστεί στο Συμβούλιο ε, για να υπερασπίσει την ε, ε, μη κατάργηση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας γιατί οι κυρώσεις σχετίζονται ε, με τιμή πρόοδο και απλώς ε, θα επιδίνουν την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Οι ε, μεταφορές κεφαλαίων από τις εθνικές αρχές είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Οποιαδήποτε λοιπόν περικαπή θα ε, είχε αντίκτυπο στον προπολογισμό τους και θα μείωνε σημαντικά την ικανότητά τους να συμμετέχουν ε, στις δημόσιες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν μια αναστολή των πληρωμών ή των ε, κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην διακοπή προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει στι περιφέρειες. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ακόμη σημείο μας βρήκε όλους ενωμένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για τις συνέργειες. 378 ε, ε, εκατομμύρια ζητάμε περισσότερο και για τις ε, συνέργειες. ναι. Υπάρχει συμφωνία, αλλά προκειμένου να γίνουν οι μεταφορέ μεταξύ των ίδιων ε, των ε, τομέων που αφορούν το Ταμείο συνοχή το 5% να μεταφερθεί, όχι πριν από το 2023 και με σεβασμό στην αρχή της εδαφικότητας, ε, έτσι ώστε τα κονδύλια που αφορούν τις περιφέρειες να γίνουν σεβαστά ως προς το κατόφλι που έχει καθοριστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ε, για το θέμα της συγχρηματοδότησης στις λιγότερο αναπτυγμένες ε, περιοχές ε, περάσαμε στο να ζητάμε από το 70% το 85% για την Νότια Ιταλία. Και Τέλος, κάτι σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι στόχοι των ταμείων θα πρέπει να συνάδουν ε, με την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, βιώσιμη ανάπτυξη, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανθεκτικότητα στους ε, ξυσμούς, ε, στις πλημμύρες και σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Εμείς αγωνιστήκαμε ε, στο ΕΤΠΑ να εισάγουμε την αρχή ε, σε ό,τι αφορά την μηδενική επιδότηση προς τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι λοιπόν θέλουμε να έχουμε μηδενικές εκπομπές άνθρακας. Δεν θα δεκτεί το Κοινοβούλιο ούτε από τους Ευρωπαίους πολίτες όμως κάποια μείωση προς τα κάτω όλων αυτών. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Σας ζητώ λοιπόν να κάνετε μια προσπάθεια και να αναφέρεστε κατευθείαν στα βασικά θέματα. Συνάδελφος Ντόιτς. Καλωσορίζουμε την κυρία Υπουργό. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το έργο της ε, Φιλανδικής Προεδρίας. Έχουμε λάβει ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την κυρία Υπουργό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε κάπως απογοητευμένοι. Ίσως ε, να μπορούσα να θέσω τρία θέματα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όταν η κυρία Υπουργό αναφέρεται στις παλιές ε, προτεραιότητες και στις νέες προτεραιότητες και ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη φράση, δηλαδή ότι η Φιλανδική Προεδρία θεωρεί σημαντικό ότι όλα έχουν τεθεί ως στόχοι στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το να υπάρχει μια εδαφική συνοχή, κοινωνική και οικονομική συνοχή και ότι αυτό θα είναι θεμελιώδες για τη Φιλανδική Προεδρία. Γιατί όταν ε, μιλάμε για ισορροπία μεταξύ νέων και παλιών προτεραιοτήτων, όταν ακούω κάτι τέτοιο, έχω την εντύπωση ότι αυτό σημαίνει ότι θέλει κάποιο να ξεχάσει τις παλιές προτεραιότητες. Δεύτερη ερώτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε μία οριζόντια συμφωνία μεταξύ των ομάδων δηλαδή ότι είναι απαράδεκτα χαμηλός ο προπολογισμό που προβλέπεται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην πρόταση της Κομισιόν και στη θέση του Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, η Φιλανδική Προεδρία θα ζητήσει αύξηση αυτού του αριθμού ή αυτό το θέμα θα αποφασιστεί μόνο και κλεισμένων το θυρών. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα κονδύλια, μεγαλύτερο αριθμό εκεί. Και τελευταία ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή των κονδυλίων για τη συνοχή. Σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση με την υποστήριξη του Συμβουλίου που ουσιαστικά θα τιμωρούσε τις χώρες εκείνες είτε στο βορρά είτε στο νότο, που έχουν αναπτυχθεί πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, όποιος είχε καλά αποτελέσματα, τώρα λαμβάνει λιγότερα χρήματα ως βραβείο. Θα αλλάξει η Φιλανδική Προεδρία αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το γεγονός ότι οι χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει καλά τα κονδύλια της συνοχής θα μπορούν να έχουν καλή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και την παρουσίασή σας κυρία Υπουργέ. Πρέπει να πω αυτής εξ αρχής ότι εγώ προσωπώ εδώ την Ουαλία, μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είναι αβέβαιη η καιρή, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως η Ιουαλία κάποια στιγμή στο μέλλον, θα μιλήσω λοιπόν επί τη βάση της συνέχισης της συμμετοχής μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η πολιτική συνοχή ήταν πολύ σημαντική για τη χώρα μου. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί, ιδιαίτερα στη Δυτική Ουαλία από, το, τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, ε, προς όφελος της ε, δικής μου εκλογικής περιφέρειας, ε, θέλω και εγώ να υποστηρίξω την αύξηση της χρηματοδότησης. Υπάρχει όμως και άλλο ένα ζήτημα. Πρέπει η οικονομία μας να αλλάξει. Πρέπει αυτό να γίνει κυρίως στις πιο φτωχές κοινωνίες. παρότι λαμβάνουμε ε, κάποια κονδύλια, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση αυτή ε, δεν θα χαθεί λόγω αλλαγής πολιτικής. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε πει ότι είμαστε κατά της πανεθνικοποίησης της πολιτικής συνοχής και νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πόσο πολύτιμο ήταν αυτό για μας πόσο κεφαλαιόδες είναι να μην χαθεί διότι η αλληλεγγύη είναι μια πολύ μεγάλη θετική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να ενισχυθεί. Η κυρία Υπουργέ, μπορείτε να μας ε, διασφαλίσετε ότι η αναφορά στο πρόγραμμά σας στην ανάγκη κοινής χρηματοδότησης στον τομέα της συνοχής ε, που θα που θα μειωθεί καθώς προχωράει η περιφερειακή συνοχή μήπως ε, σημαίνει επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής. Αν όχι να μας το πείτε. Σε ό,τι αφορά τώρα την απανθρακοποίηση ε, ε, είναι 25% η πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο προτείνει 30%. Εσείς ποια είναι η δική σας θέση από αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεχουμέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στην πρόταση μείωσης ε, του προπολογισμού σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία ε, απασχόληση των νέων. Είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Προέρχομαι από την Ισπανία, όπως ξέρετε, το μέσο ποσοστό ανεργίας για τους νέους είναι γύρω στο 34%. Ε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε επί Ισπανικής Προεδρίας ε, ε, με κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας. Τότε ε, ήταν πολύ πιο υψηλά τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον πλέον επιτυχή τρόπο. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μία από τις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους νέους που ψάχνουν θέση εργασίας, που θέλουν να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους, που θέλουν να έχουν την ευκαιρία ε, να ε, βελτιώσουν την κατάστασή τους στα κράτη-μέλη στα οποία ζουν. Εάν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε τις ανισότητες, η ανισότητα μειώνεται δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης δημιουργώντας ε, πλούτο για να μπορούν οι νέοι στις δικές τους χώρες ε, να πάρουν τις πρωτοβουλίες που θέλουν να πάρουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην μειωθεί ο προπολογισμό αυτός, ε, να έχουμε κατά νου τους νέους και να ξανασκεφτούμε ποιοι είναι τελικά οι στόχοι και ποια είναι οι χρήσει αυτού του προπολογισμού αλλά σε κανένα περίπτωση δεν πρέπει να μειωθεί. Πρέπει να βρούμε το πιο αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών, εάν θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία των νέων και να του δώσουμε ευκαιρίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Μαρτέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία. Υπουργέ, Εσεί προέρχεται από μια χώρα στο βορρά και όπω και δική μου χώρα που είναι στο νότο έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά προκλήσεων. Έχουμε κοινέ προκλήσει, ε, παραδείγματο χάρη, η μείωση του πληθυσμού και άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Μίλησατε για την ε, περιφερειά σας, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας. Εγώ προέρχομαι από την ε, Καστίγια Λαμάντσα. Εκεί υπάρχουν κάποιες κομματίε όπως η Κουένκα, η Σιουδάδ Δρεάλ, όπου τα τελευταία χρόνια πάνω από το 90% των δήμων έχουν ε, χάσει τον πληθυσμό τους και συνεχώς χάνουν σε πληθυσμό και υπάρχουν πάρα πολλοί πυρήνες, υπάρχουν κάποια χωριά, έχουμε μόνο, παραδείγματος χάρη, 8 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Είναι πάρα πολύ μικρή η πυκνότητα του πληθυσμού και είναι πάρα πολύ σημαντικές και προκλήσεις. Έχουμε χαμηλή ε, γενετικότητα, έλλειψη βασικών πόρων για την απασχόληση, για την υγεία και έχουμε και πολύ χαμηλή απασχολησιμότητα. Εμένα μου άρεσε πολύ που εσείς αναφέρατε ρητός την πρόκληση της δημογραφίας ως μια πρόκληση για το μέλλον. Όμως πολλά πρέπει να γίνουν. Σε αυτό το κοινοβούλιο σημειώσαμε μεγάλη προόδο. Έχουμε εγκρίνει σημαντικές εκθέσεις που επέτρεπαν με οριζόντιο τρόπο να προσεγγιστεί το θέμα της μείωσης του πληθυσμού στις πολιτικές συνοχής. Όμως εγώ θα ήθελα να τονιστεί ακόμη περισσότερο να μας πείτε πείτε ποιες πολιτικές εσείς θέλετε να υλοποιήσετε ε, προκειμένου ε, να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σημαντική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τα επόμενα έτη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ward. Επίσης έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από άκουσα από τη Φιλανδική Προεδρία. Και μαζί με την Jill Evans είχα και εγώ την ευκαιρία να κάνω μία επίσκεψη μελέτη στη Φιλανδία τον Ιανουάριο, πριν 18 μήνες περίπου. Εκεί εξετάσαμε το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ε, και της επιχειρηματικότητας και το ψηφιακό θεματολόγιο. Γνωρίζω ότι η Φιλανδία έχει ηγετική θέση σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική της πολιτική. Ουσιαστικά ε, άκουσα να μιλάτε για επαφές μεταξύ των ανθρώπων και με εξέπληξε θετικά αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε για την περιφερειακή πολιτική και τα διάφορα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Εγώ ενδιαφέρομαι κυρίως για τον πολιτισμό και την ε, παιδεία. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν εν μέρη υπεύθυνη για ένα φάκελο για την κοινωνική συνοχή και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Η ακρόση που οργανώσαμε σε αυτή την επιτροπή χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα των πρακτικών ε, από μια οργάνωση για τις τέχνες ε, που εργάζεται σε ένα πλαίσιο κοινωνικής στέγασης ε, στην ε, βορειοδυτική Αγγλία, σε μια πολύ φτωχή περιοχή. Οι τέχνες ε, και ο πολιτισμός διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στο να διευκολύνουμε την επαφή μεταξύ των ανθρώπων και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και αυτό δεν αποκλειστήκε αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού. Γι' αυτό μου άρεσε που αναφερθήκατε στην επαφή μεταξύ των ανθρώπων θα ήθελα όμως ε, να μας πείτε λίγο περισσότερο για το πώς βλέπετε εσείς ε, η παιδεία και οι τέχνες να τεθούν περισσότερο στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτή την πολιτική στο έργο των διάφορων επιτροπών και των τομέων πολιτικής. Ευχαριστώ. Και τώρα Κυρία Πεκάρινεν από τη Φιλανδία. Ο κύριος Πεκάρινεν, παρακαλώ, έχετε στήσει το λόγο. Φιλανδία. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ, που σας συναντώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι Φιλανδός, το ξέρετε. Και έτσι έχω μια πολύ πολύ απλή ερώτηση. Την εξή. Πιστεύετε ότι στη διάρκεια της φιλανδικής προεδρίας θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτή την τόσο βαριά γραφειοκρατία που ε, συνεπάγεται η διαχείριση σε πρακτικούς και καθημερινούς όρους της πολιτικής συνοχής. Έχω εγώ τελέσει και υπουργό, έχω λάβει αποφάσεις, είχα ευθύνη αυτών των φακέλων και πρέπει να πω ότι η διαδικασία είναι η εξής. Η Επιτροπή δίνει κατευθύνσεις, προσανατολισμούς δηλαδή για την προσεχή ε, προγραμματική περίοδο, τι θα πρέπει να γίνει, που δίνεται έμφαση. Μετά πάνε τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν τις ιδέες, μετά τα στέλνουν στις περιφέρειες με τους προσανατολισμούς τους, μετά οι περιφέρειες προσπαθούν να στήσουν τα δικά τους τα προγράμματα σε επικοινωνία με τα Υπουργεία. Μετά γίνεται αυτό το πηγενέλα με το feedback που πρέπει να δοθεί από την περιφέρεια στο κεντρικό κράτος κτλ. Μετά οι τοπικές αρχές θα ξαναμιλήσουν με το τον Υπουργό, μετά ο Υπουργός θα ξαναγυρίσει να μιλήσει με τους εκπροσώπους Επιτροπής. Ε, πάνω κάτω δεξιά αριστερά ε, ένα πήγαινε ένα γραφειοκρατικό τερατόδε, το οποίο τελικά πολύ λίγο αντιστοιχεί ως επιβάρυνση με το ποσό που τελικά ορισμένες περιφέρειες τουλάχιστον θα πάρουν. Δεν είναι καθόλου λογικό όλο αυτό. Για χρόνια προσπαθήσαμε να περιορίσουμε αυτή τη γραφειοκρατία. Έχω όμως την ε, εντύπωση ότι μόνο πληθαίνει το χαρτομάνι και η γραφειοκρατία. Θα κάνετε κάτι, πιστεύετε ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πόλακ. Ο κύριος Πόλακ έχει σπίσει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιες ε, χώρες όπου είναι δύσκολο ακόμα και να εξασφαλίσουν οι πολίτες πρόσβαση σε, πόσιμο νερό στον 21ο αιώνα. Και όμως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες δεν έχουν ούτε κατάλληλη αποχέτευση, ούτε πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή δρόμους ε, σε επίπεδο ικανοποιητικό. Μιλούμε για περιορισμό των διαφορών μεταξύ των περιφερειών. Ναι, Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ο καθένας μας πρέπει να καταβάλει, δηλαδή, ε, το μέγιστο των προσπαθειών του για να εξασφαλίσει ένα καλό επίπεδο για όλες τις περιφέρειες. Και πρέπει, πιστεύω, να εξασφαλίσουμε πάνω απ' όλα οι λιγότερο πλούσιες περιφέρειες να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε να προσφέρουν στους πολίτες τους τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης που αξίζουν πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης, απόκτηση δεξιοτήτων με την εκπαίδευση, την κατάρτιση κτλ. Αυτά δεν τα αναφέρατε καθόλου στις προτάσεις σας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια για το εκείς Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριο κύριος Κιμπρούκλος, παρακαλώ. Έχετε το λόγο πολύ για το λόγο κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ. Ε, προέρχομαι, είμαι ένας νέος άνθρωπος, ε, προέρχομαι από μια χώρα η οποία δυστυχώς ε, οι, διάφορες, ε, οι διάφοροι πληθυσμοί οι οποίοι θεωρούνται περιθωριοποιημένοι έχουν ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Ε, θα συμφωνήσω απόλυτα με την συνάδελφό μου προηγουμένως. Ε, όμως είμαστε και μια χώρα η Ελλάδα που μπαίνει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και είμαι σίγουρος ότι γρήγορα θα κάνει την ε, έκπληξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο για να, βγούμε από αυτή την ε, χρόνια ύφεση που βρεθήκαμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι περιφέρειές μας όπως η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως και η περιφέρεια της Υπήρου δυστυχώς πρωτεύουν σε, αυτήν σε αυτό το, τον αγώνα της ανεργίας. Ε, Ιδίω για τις νέους και τις γυναίκες. Τα νησιά επίσης, επίσης πλήττονται από το γνωστό ε, στην Ελλάδα brain drain ε, και δέχονται πολλές προκλήσεις. Ε, και αναρωτιέμαι, τι προβλέπετε λοιπόν να κάνετε ε, για τις περιφέρειες με μεγάλη ανεργία, ειδικά σε, στις ειδικές ομάδες, νέους, γυναίκες, ε, ανάπηρους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Et pour une dernière prise de parole, Ευχαριστώ τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Η καινοτομία ε, και η έρευνα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την απασχόληση, την ποιοτική, για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Πρέπει είναι σημαντικό να υπάρχουν ε, τα απαραίτητα κονδύλια για να υποστηρίξουν τι μικρέ επιχειρήσει, του επιχειρηματίε. Είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι, καθώ και το θέμα τη ψηφιακή μετάβαση, θα πρέπει το ευρυζωνικό να φτάσει σε όλε τι περιοχέ τη Ευρώπη και στην Ήπεθρο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είναι ε, η απερίμωση. Δεν πρέπει κανεί να μείνει μόνο, του, κανείς να μείνει πίσω, λέει η κυρία Σόλη Πέρεθ. Ε, δεν ξέρω εάν η καινοτομία για εσά στι περιφέρειες τη ευρωπη είναι προτεραιότητα τη Φιλανδικής προεδρία. σα ζητάω λοιπόν, ποια, ρωτάω, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θέλετε να πάρετε και να εξασφαλίσετε ότι διαπραγματεύσει οι και διαπραγματεύσει ε, για τα ταμεία ε, θα δουν την καινοτομία στο κέντρο των συζητήσεων ε, και των, της πολιτικής συνοχής. ευχαριστώ και καλή τύχη για την Προεδρία σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Οι πολυέρθμες ερωτήσεις μας δείχνουν πως μεγάλη προσοχή δίνει η δική μας Επιτροπή στο θέμα της συνοχής ε, και στην Προεδρία σας. Ελπίζουμε να απαντήσετε συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Αριμού για το Interreg. Και για το θέμα της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής. Στην περίπτωση του Interreg, εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει ένας τριμερής διάλογος για τον κανονισμό Interreg, όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες του κανονισμού αυτού και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αποκλήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το πώς πρέπει να εξελιχθεί αυτός ο κανονισμός Interreg. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή έκβαση σε αυτό το φάκελο. Επίσης, Τέθηκε μια ερώτηση για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και αναφέρεστε πάρα πολύ εσείς σε αυτό, είναι και λογικό. Βεβαίως το θέμα της χρηματοδότησης πάντοτε ξυπνά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Σαριμών ρώτησε σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και αν θα έπρεπε αυτή η χρηματοδότηση να αυξηθεί. Εγώ πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε προς ε, τα που θα κινηθεί η συζήτηση για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των προγραμμάτων και όλων αυτών των πολιτικών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Φιλανδία ως Προεδρία δεσμεύεται έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση να προχωρήσουν. Θέλουμε να πετύχουμε μία συμφωνία πριν από τα τέλη του έτους. Σε αυτό δεσμευόμαστε. Τώρα, σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχή και για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις ανισότητες ανάπτυξης μεταξύ των διάφορων περιφερειών, η κυρία Μαρτίνη, η κυρία Εύανς επίσης αναφέρθηκαν σε αυτά τα θέματα. Ο έσχατος στόχος θα πρέπει να είναι το χάσμα να μειωθεί μεταξύ των διάφορων περιφερειών και σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ η πολιτική συνοχής. Είναι όρατα τα αποτελέσματα. Επομένως, πρέπει να πούμε ότι η πολιτική συνοχής παρουσιάζει αποτελέσματα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Έχει βοηθήσει στο να μειωθούν ε, οι αναπτυξιακέ ανισότητε μεταξύ των διάφορων περιφερειών. Βέβαια, συνεχίζουν να υπάρχουν ανισότητε, το είδαμε και στη συζήτηση. Όπω και να έχει, η πολιτική συνοχή μπορεί να συνεχίσει να είναι μια πολιτική που παρουσιάζει αυτά αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η πολιτική. Το είδαμε, παραδείγματο χάρη, και στην ε, έκθεση κοινωνικής ανάπτυξης του 2017 ε, και είδαμε πώς κοινωνικά η πολιτική συνοχής και σε άλλους τομείς παρουσίασε θετικά αποτελέσματα. Είναι βέβαιο ότι πάντοτε υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε κάποιες περιοχές, όπως το χάρη το θέμα της μείωσης του πληθυσμού. Ο κύριος Ντόιτς έθεσε μια ερώτηση για τις νέες προτεραιότητες έναντι των παραδοσιακών πολιτικών και πώς θα βρούμε μία ισορροπία μεταξύ των δύο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να βρεθεί αυτή η ισορροπία και εργαζόμαστε για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Όμως, βεβαίως, πάντοτε πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Αυτό είναι σαφές. Αυτό έχει καθιερωθεί και στις συνθήκες. Γιατί η εξέβρεση με, της ισορροπίας μεταξύ παλιών και νέων πολιτικών ε, πρέπει να γίνει, όμως πάντοτε θα πρέπει να έχουμε κατά νου ποιος είναι ο κοινός μας στόχος. Σε ό,τι αφορά τώρα την κοινωνική προοπτική, η κυρία Γουόρτ έθεσε το κοινωνικό ζήτημα και δεν ήταν η μόνη. Μίλησε όχι μόνο για την κοινωνική διάσταση, αλλά και για την ε, συγκεκριμένη περίπτωση των νέων. Η Φιλανδική Προεδρία θεωρεί ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να τεθούν ε, σε ευρεία βάση. Η αντιγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμβαδίζει με την κοινωνική ένταξη. Παραδείγματο χάρη, οι σχέσεις μεταξύ των γενεών, η κοινωνική ευημερία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον. Η Φιλανδία θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει το κοινωνικό συστός. Εδώ ο κοινωνικό πυλώνα θα αποτελεί ένα στοιχείο που θα βαρύνει ιδιαίτερα στην εντολή του Συμβουλίου και σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος ε, Πιέιτ Κάρινεν ρώτησε για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Η διαχείριση της πολιτικής συνοχής ε, δεν θα πρέπει να ε, σημαίνει ότι είναι υπερβολικό το διοικητικό άχθος. Και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε απλούστευση της διαχείρισης. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποια βήματα Προ την μείωση τη γραφειοκρατίας ε, προκειμένου να πλουστευτεί η διαδικασία και εμεί υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο σύντομου κανονισμού. Δεν ε, χρειάζεται μία νομοθετική πράξη, από τη μία νομοθετική πράξη στην άλλη να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες διατάξεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτή η επανάληψη. Θα έπρεπε επίσης ε, να μειώνουμε και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη των προγραμμάτων, έτσι ώστε Μάλλον εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να απλουστευτούν τα νομοθετήματα και αυτό θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη ευελιξία κατά την άποψή μας. Η κυρία Σολής Πέρες έθεσε ένα ερώτημα που αφορά το πρόγραμμα εργασίας μας, το οποίο βασίζεται πολύ στις νέες τεχνολογίες, στις νέες τεχνολογίες περί στην καινοτομία. Θεωρούμε ότι η στρατηγική, η ευφυή στρατηγική εξειδικευσή ε, θα μπορέσει επίσης να οδηγήσει στην καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, να μπορούν οι περιφέρειες να αναπτύξουν, να αναπτυχθούν στον τομέα που είναι καλύτερες. Νομίζω ότι αξίζει να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Προσπάθησα λοιπόν να απαντήσω στις ερωτήσεις που σημείωσα. Προσπάθησα να απαντήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου. Φυσικά συνεχίζω να είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω και γραπτός αν ε, θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαι στην διάθεσή σας για να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτά τα ζητήματα που, όπως είπα, είναι ζωτικά για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση μαζί σας, να ακούω τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις αμφιβολίες σας. Προσωπικά είμαι πεπισμένη ότι η πολιτική συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης ε, θα προχωρήσουν γιατί είναι σε καλά χέρια. Έχουμε να λάβουμε πάρα πολλές δύσκολες αποφάσεις, πολύπλοκες αποφάσεις. Μεταξύ αυτών πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτά τα θέματα για αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν ίσως κάποιες επώδυνες αποφάσεις ε, σε όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής. Ε, θα πρέπει όλοι μας να εργαστούμε για να μπορέσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις και να λάβουμε τις καλύτερες αποφάσεις έτσι ώστε να συνεχίσει με φυή τρόπο και με δίκαιο τρόπο να αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένω, είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω μαζί σας όποτε το κρίνετε χρήσιμο και η Φιλανδία δεσμεύεται στην Προεδρία της να προωθήσει τη δέσμη μέτρων για τη συνοχή. Εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των συναδέλφων και ελπίζω από την συνάντηση αυτή να πάρετε μαζί σας το πολύ υψηλό φρόνημα της Επιτροπής μας. Σκοπεύουμε να κάνουμε να εισακουστούν οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην κλείσει το δρόμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο δρόμο για την αναζήτηση μιας συμφωνίας για το πολιτές νοσονομικό πλαίσιο, μια συμφωνία και για τις παραδοσιακές ε, πολιτικές και πολιτική και κυρίω πολιτική της συνοχής. Και βεβαίως το Κοινοβούλιο θα υψώσει το ανάστημα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, είμαι βεβαίως. Δεύτερον, πιστεύω πως η Προεδρία σας θα πρέπει να αποστείλει ένα θετικό μήνυμα που θα ευνοήσει συνομιλίες που θα έχουμε σύντομα και τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Η οργάνωση ενός άτυπου συμβουλίου για το θέμα έχει μεγάλη σημασία για μας. Ιδάλλως, αυτό θα σημάνει μία ρήξη και δεν θα είναι βέβαια καθόλου θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και τη συμμετοχή σας και σας δίνω ραντεβού πολύ σύντομα, ούτως ή άλλως είμαστε καταδικασμένοι να ξανασυναντιόμαστε στο επόμενο εξάμεινο τακτικά. Nous poursuivons notre réunion. Celles et ceux qui quittent la salle, je vous remercie de le faire. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ όποιο είναι να αποχωρήσει ήσυχα για να συνεχίσουμε. Merci de quitter la salle en silence pour que nous puissions... Ναι, παρακαλώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε την ημερήσια μας διάταξη. <laughs> λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μα. Σήμερα το πρωί δεχτήκατε τροποποίηση τη σημερινή διάταξη για να δούμε σήμερα, για να δούμε τώρα μάλλον το σημείο 4. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρία των συντονιστών σήμερα το πρωί, επιβεβαιώθηκε ότι οι συντονιστέ θέλουν η Κομισιόν να ακολουθήσει τη σύνοδο πρακτική, ε, τη σύνηθη πρακτική σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαδικασία. Ο πρόεδρος λοιπόν θα είναι εισηγητή για τη συνεισφορά της δική μα επιτροπής, τη επιτροπή Ρέτζη, στην δημοσιονομική διαδικασία ε, για το 2020. Ο πρόεδρος επιφορτίζεται επίση με την κύρωση οποιασδήποτε μείωση εισαγάγει το Συμβούλιο στο το σχέδιο του, της Κομισιόν και να προτείνει προτάσεις ε, δράσεων πιλωτικών και προπαρασκευαστικών, προπαρασκευαστικών μέτρων που αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης αξιολόγησης από την Επιτροπή. Εάν θέλουν να υποβάλουν οι βουλευτές άλλες τροπολογίες ή να προτείνουν άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα και πιλωτικές δράσεις θα πρέπει να το πράξουν απευθεία στην Επιτροπή Προπολογισμού, στη Δημοσιονομική Επιτροπή, ενημερώνοντα ε, βέβαια και τον πρόεδρο της επιτροπή Ρέτζη. Ο πρόεδρο λοιπόν θα προετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότηση για την πρόταση ψηφίσματο ε, για τον προπολογισμό. Θα υποβληθεί 3 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Ρέτζη ε, αυτό το σχέδιο και ελπίζουμε να ψηφιστεί στη συνεδρίασή μας 2 και 3 Οκτωβρίου. Έως τώρα οι βουλευτές έχουν προτείνει 12 πιλωτικές δράσεις και προπαρασκευαστικά μέτρα που αποτελούν αντικείμενο μιας πρώτης αξιολόγησης από την Επιτροπή. Μία εξ αυτών απεσύρθη η 11 που απομένουν θα υποβληθούν εκ μέρους, μου, εκ μέρους της Επιτροπής μας από εμένα. Επίσης, στις 10 Ιουλίου το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Το Συμβούλιο επέφερε κάποιες λίγες τροποποιήσεις στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τίτλο 13, περιφερειακή πολιτική και αστική πολιτική, που είναι και το θέμα που μας απασχολεί, η... το Συμβούλιο έχει μειώσει ε, τις δεσμεύσεις για τις μαστονομικές γραμμές που έχουν να κάνουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και την τεχνική συνδρομή και τις καινοτόμες δράσεις και τις πληρωμές για την γραμμή τη δημοσιονομική για την αποσχόληση των νέων. Εγώ λοιπόν θα υποβάλω τροπολογίες για να ακυρωθούν αυτές οι μειώσεις που προτείνει το Συμβούλιο. Ε, μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτήν την σημαντική πτυχή. Το είδαμε άλλωστε και στη συζήτηση που μόλις είχαμε με την Υπουργό τα δημοσιονομικά ζητήματα είναι στην καρδιά ε, της συζήτησης, διότι μόνο με τα, κατάλληλα κονδύλια μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνοχή. Θα δώσω λοιπόν, τώρα λοιπόν το λόγο στους σκιώδης συζητητές για το ΕΛΚ είναι κάποιος εδώ, σκιώδης συζητητής. Δεν υπάρχει ε, σκιώδης του ΕΛΚ εδώ από τους σοσιαλιστές. Ναι, προσωπεί τον κύριο Πέκουλα. Υπάρχει λοιπόν σκιώδης συγητής. Ναι. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου όμως ο μιλητής και δεν τον ακούμε και δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Ναι. Όντω, αντικαστώ τον κύριο Πίκολα που μου ζήτησε να διαβάσω ε, αυτά που έχει να σας πει. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην απογευματινή συνεδρίαση ε, επειδή είχα κάτι άλλο στο πρόγραμμά μου ε, την ίδια ώρα. Μας περιμένει πολλή δουλειά το φθινόπωρο. Θα, ο κ. Πέκολα συμφωνεί με την διαδικασία που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών. Λάβαμε 7 προτάσεις από τους συνοδέλφους της προηγούμενης θητείας, 4 πιλωτικά προγράμματα και τρεις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις. Αναμένουμε ακόμα την αξιολόγηση της τελευταίας πρότασης που, υπέβαλε, που υπέβαλαν οι νέοι συναδέλφοι. Συνάδελφοι, από τον κύριο Κοτσολίνο θα συνεχιστεί η διαδικασία το Σεπτέμβριο, θα υποβληθούν τροπολογίες προς τον προπολογισμό και θα, ψηφιστούν. Γενικότερα, για το θέμα του προπολογισμού δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ε, που θα οδηγήσει το Brexit, ιδιαίτερα μετά και τα σημερινά νέα. Ε, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο προπολογισμό πάντω για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σχετική πολιτική και ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή, που είναι κεφαλαιόδε μέρο τη ε, περιφερειακή πολιτική. Ε, εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία και καλέ διακοπέ σε όλου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Αντρέι Νοβάκοφ μια σύντομη διευκρίνηση επειδή η απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαδικασία υπάρχει πριν από μία ώρα περίπου, υπάρχει μια έκκληση για το ποιος ενδιαφέρεται για ως συγκητής στην ομάδα μας. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση, ε, αλλά θα την έχουμε πολύ σύντομα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ως συγκητής από το ΕΛΚ εδώ. Μάλιστα, πολύ ωραία για την ομάδα Renew. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι, ορίστηκα εγώ σχεδόν συζητητής, ε, θα το συζητήσω όμως και με τους συναδέλφους ε, και θα υποβάλουμε συγκεκριμένες ε, τροπολογίες το Σεπτέμβριο. Δεν αναμένουμε πάντως να προσθέσουμε νέα στοιχεία σε παιδοπιλωτικών προγραμμάτων. Ενδεχομένως να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες το Σεπτέμβριο με βάση και το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε για τους πράσινους, κυρία Αγγής. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε να δώσουμε εντολή στον Πρόεδρο. Αλλά ως προς το περιεχόμενο θέλω να το σχολιάσω τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο γιατί οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ. Αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ χαμηλή η στόχη. Έχουμε και ένα πιλωτικό σχέδιο για το climate proofing και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να δώσουμε πραγματικό αγώνα κατά της κλιματικής συλλογή. Αυτό θέλαμε να σας παρουσιάσουμε για τις διαπραγματεύσεις. De prise de parole. Ζητά άλλο το λόγο από κάποια άλλη ομάδα. Όχι. Πιστεύω ότι έχει πλαισιωθεί η διαδικασία. Θα ήθελα να διορίσετε τους κοιόδης εισηγητές έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και βέβαια ως εισηγητής είμαι στη διάθεσή σας και όπως σας είπα θα καταγράψω τα αιτήματα. Σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε στα πλαίσια της συνεδρίας των συντονιστών, να έχετε λάβει και τις αποφάσεις τους. Σας ζητώ να εγκρίνετε τις αποφάσεις ε, των συντονιστών. Πολύ ωραία. Άλλα θέματα που θέλουν να θέσουν ε, οι βουλευτές. Κάποια θέματα στα οποία θέλετε να αναφερθείτε. Όχι. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, σας δίνω ραντεβού για την ε, επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, στις 3 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί, στις Βρυξέλλες. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για την ποιότητα των ερωτήσεων που τέθηκαν στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα.